με αυτή. Σύμφωνα με την Περισσία Διάταξη, περνάμε τώρα στην κοινή συζήτηση για τη δήλωση τη Κομισιόν και του Συμβουλίου για τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση στο και τη σύσταση Αλόη Πέτολε για τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση στο Καταρχήν θα δώσω το λόγο με μεγάλη χαρά στην τέο συνάδελφο. Πρόεδρο του Συμβουλίου, κυρία Μάνιστρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Επίτροπε, κύριε Σιγητά, κύριε Πέτρελε. Είμαι ευτυχή που μπορώ να συζητήσω σήμερα το απόγευμα τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ενώσεω με το Τατζικιστάν. Είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε τη σχέση με αυτή τη χώρα υπογράφοντας αυτή τη ε, συμφωνία εταιρική σχέσεως και συνεργασίας. Το κοινοβούλιο μας πάντα έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα θέματα. Το Φεβρουάριο του 2008 στο ψήφισμά σας για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσης για την Κεντρική Ασία ζητήσατε κάτι μελη να κυρώσουν γρήγορα τη συμφωνία ε, συνεργασίας και εταιρική σχέσεως και επιβεβαιώσατε τις προθέσεις του Κοινοβουλίου κάνοντας το αυτό, επικυρώνοντας αυτή τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία λοιπόν επικυρώνεται και υπάρχει επιθυμία να προχωρήσουμε και να κάνουμε και τα επόμενα βήματα, ώστε η συμφωνία αυτή να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν και ελπίζουμε πριν το τέλος του έτους. Τότε θα στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Τατζικιστάν. Κυρίες και κύριοι, το Τατζικιστάν είναι σημαντική συνιστόσα της στρατηγικής μας για την Κεντρική Ασία. Ε, είναι χώρα απομονωμένη, πολύ δύσκολο να φτάσει κανεί, είναι από τι στοχότερε, έχει σύνορα τα οποία δεν φυλάσσονται καλώ με το Αφγανιστάν και περνάνε πολλά ναρκωτικά από εκεί. Είναι μια πύλη ε, για ακρεφνεί Ισλαμιστέ και γι' αυτό μα ενδιαφέρει η υποστήριξη του Τατζικιστάν και προ όφελο τη χώρα και για να λύσουμε κοινά προβλήματα. Ήδη είχα κάποιε επαφέ. Η Σουηδική Προεδρία έστειλε ομάδα υψηλού επίπεδου στην περιοχή τον Ιούλιο και έγινε διπουργική διάσκεψη για την Κεντρική Ασία στι Βρυξέλλες ΧΤΕ. Το Τατζικιστάν είναι μία από τις λίγε χώρες στην περιοχή την Ανατολική της Ευρωπαϊκής Ενώσης με την οποία δεν έχουμε μία ξεκάθαρη συμφωνία μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να αντιμετωπίσουμε τα προαναφερθέντα θέματα θα πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο για διμερείς ε, σχέσει. Ε, οι διευθετήσει για πολιτικό διάλογο και πρακτική συνεργασία με το Τζικιστάν πρέπει να βελτιωθούν για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τι προκλήσει τη περιοχή. Αυτή η συμφωνία εταιρική σχέσεω και συνεργασία θα μα επιτρέψει μια πιο δομημένη προσέγγιση για τη συζήτηση κοινών θεμάτων όπω είναι το κάτω δικαίου, καταπολέμηση των αθρεμπορίων ναρκωτικών, καταπολέμηση του οργανωμένου κατά καταπολέμηση τη τρομοκρατία και του ε, θρησκευτικού φονταμεταλισμού. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε θέματα όπω είναι η δημοκρατία, η καλή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή. Βεβαίω ε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά δεν είναι εύκολα και γι' αυτό με μεγάλη χαρά βλέπουμε ένα δομημένο διάλογο με το Τατζικιστάν που δημιουργείται και αυτό θα μας επιτρέψει μια σωστή συζήτηση με αυτού τους ανθρώπους. Και αυτός ο διάλογος θα γίνει στον Τουσάμπε στις 23 ε, Δεκεμβρίου. Πρέπει να βοηθήσουμε το Τζικιστάν να ολοκληρώσει τι μεταρρυθμίσει. Πολύ συχνά οι εξελίξει εκεί είναι ανησυχητικέ. Θέλουμε να υπάρξουν μεγαλύτερες δημοκρατικές προοπτικέ για τη χώρα, όπως το δικαίωμα του συνεταιρίζεσαι, το δικαίωμα της, της, ε, ε, την ε, το κάτος δικαίου θα πρέπει το κράτο δικαίου να ισχύσει και να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και τρομοκρατία. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Και αυτό είναι ένας τρόπος ε, να αποφευθούν πολιτισμικές συγκρούσει ή εθνοτικέ συγκρούσει. Ανησυχούμε πολύ για την διαφθορά που υπάρχει στη χώρα που εμποδίζει την ανάπτυξη του Τατζικιστάν και εμποδίζει και τη χορήγηση δωρεών. Ε, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι επιχειρήματα έχουμε για να πείσουμε τις αρχές της χώρας να αντιμετωπίσουν το ταχύτερο δυνατό αυτό το πρόβλημα της διαφθοράς. Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορούμε να κλείσουμε το μάτι όσον αφορά τη διαμετακόμιση ε, των ναρκωτικών που περνάνε από το Ταζικιστάν και εκτίθεται σε ριζοσπαστικά κινήματα και το διεθνέ οργανωμένο έγκλημα η χώρα. Θα πρέπει να αυξήσουμε την υποστήριξή μα για το Τατζικιστάν, να μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει αυτέ τι δραστηριότητε. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και άλλε εναλλακτικέ μορφέ εισοδήματο για τη χώρα, εσόδων για τη χώρα. Αυτό ταιριάζει και με τι υποχρεώσει που έχουμε αναλάβει στο Αφγανιστάν και την προσπάθεια που καταβάλουμε να σταθεροποιήσουμε αυτή τη χώρα. Και καλωσορίζουμε το ενδιαφέρον του Τατζικιστάν που θέλει να συνεργαστεί μαζί μα και να συμβάλλει σε αυτέ τι προσπάθειε. Το Τατζικιστάν έδειξε επικοδομητική στάση, ανοιχτή στάση στη συζήτηση των κοινών προβλημάτων και προκλήσεων και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Αυτός ο διάλογος είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Τώρα που θέλουμε να βοηθήσουμε τον Τατζικιστάν, θέλουμε να συνεργαστούμε ε, με τις γειτονικές του χώρες και θέλουμε να βρούμε λύσεις για κατεμπήγοντα περίπλοκα ε, περιφερειακά προβλήματα όπως τη διαχείριση των υδάτων, η αλλαγή του κλίματος και άλλα συναφή. Θα είναι πολύ χρήσιμο λοιπόν να συνεργαστούμε με το Τζικιστάν για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτή η συμφωνία θα μα δώσει ένα πλαίσιο εντό του οποίου θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τι διμερεί μα σχέσει και ούτω τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε στην επίτευξη των γενικότερων στόχων στρατηγική μα στην Κεντρική Ασία. Και γι' αυτό καλό το Κοινοβούλιο να συμφωνήσει με αυτή την συμφωνία, ούτω ώστε να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Το λόγο έχει ξενομιδότηση της Κομισιόν η Επιτροπής κυρία Φέρε Βάλλον. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, καταρχήν επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτερλε για την θαυμάσια του έκθεση και για το ψήφισμα το οποίο αναλύει πάρα πολύ καλά την κατάσταση στο Τατζικιστάν και προετοιμάζει δηλώσει και συστάσει που μπορώ να υποστηρίξω. Από τότε που εθετήθηκε η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ασία από τον Ιούνιο του 2007, οι σχέσει μα με όλε τι χώρε τη Κεντρική ε, Ασία έχουν ευαθυνθεί προ όφελο και των μεν και των δε. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ μα έχει αυξηθεί και τώρα καταναούν όλοι τα ωφέλη από καλύτερη συνεργασία σε θέματα ασφάλεια παιδεία, ε, διακυβέρνηση και διαφοροποίηση των πηγών ενεργείας. Η στρατηγική αυτή προωθεί ένα νέο είδη εταιρική σχέση με τις ε, δημοκρατίες αυτή τη Κεντρική Ασία. Βέβαια, αυτή η στρατηγική βασίζεται σε διαφοροποιημένες διμερείς σχέσεις που αντικατοπτρίζουν διαφορετικές ε, προοπτικέ ε, και προσπάθειες των ε, κρατών αυτών. Ξέρετε ότι η συνεργασία με το Τατζικιστάν αυτή τη στιγμή ελέγχεται από τη Συμφωνία Εμπορίου και συνεργασία που είχε συναυτεί το 1989 με την Σοβιετική Ένωση και υποστηρίχθηκε από το 1994 από το Τατζικιστάν. Δεν αντικατοπτρίζει δηλαδή πλήρως Τη ε, φιλοδοξία μας μέσα στα πλαίσια στρατηγικής για την Κεντρική Ασία, ούτε υποστηρίζει εκείνες τι σχέσει που αυτή τη στιγμή αναζητούμε με το Τατζικιστά. Η έγκριση από μέρους της νέας ε, συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τατζικιστάν που έχετε αυτή τη στιγμή ενώπιον σας να εξετάσετε θα μας προχωρήσει και θα μας επιτρέψει να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με τη χώρα αυτή. Το Τατζικιστάν σήμερα αντιμετωπίζει, όπως ελέγχθη, τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Είναι σημαντικό και προ όφελο των Ευρωπαίων το Τατζικιστάν να καταφέρει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες αυτές, γιατί πρόκειται για μια χώρα η οποία έχει περίπου 1500 χιλιόμετρα σύνορα με το Αφγανιστάν και βρίσκεται πολύ καλά στην ε, ε, κοιλάδα του Σπάτ με το Πακιστάν. Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε ότι εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα λόγω της, ε, του ότι είναι τόσο σε αυτοί οι ε, πυρήνες τόσο προβληματικοί. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη αστάθεια στη χώρα ένα κύριο στοιχείο της, ε, του λόγου γιατί το Τατζικστάν είναι τόσο ευάλωτο είναι η αδύναμη οικονομία του γιατί ε, πλήγησαν από τη μείωση των τιμών για αλουμίνιο και για χαλκό λόγω της μείωσης της οικονομικής ε, ανάπτυξης παγκόσμια. Αυτό οδήγησε σε ε, τεράστια ποσοστά μείωσης των εσόδων της χώρας και γι' αυτό ίσως αυξάνονται επίπεδα ένδυας και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που είναι πολύ επισφαλής θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνική επανάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη χώρα αυτή, πράγμα που ήταν και το επίκεντρο των προσπαθειών του κυρίου Μπορέ του ειδικού αποσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δικών μου επισκέψεων την Άνοιξη. Υπάρχει πρόοδος, θα πρέπει όπως πολλά περισσότερα να γίνουν διευκρίνησε η κυβέρνηση ότι ε, προτίθεται να επιβάλλει μέτρα που θα βοηθήσουν την κοινωνική ευμάρεια, την υγεία, την παιδεία, να αντιμετωπίσει την, <clears throat> ε, τις δωροδοκίες και είναι σημαντικό που δημιουργήθηκε η θέση ενός ε, διαμεσολαβητή, ενός συνηγόρου του πολίτη, πράγμα που θα μας βοηθήσει στις μελλοντικές ε, συζητήσεις στις 23 Σεπτεμβρίου με τη χώρα αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρόταση είναι αργή, αλλά ελπίζουμε ότι οι συστάσεις μιας πρόσφατης ε, ε, συνάντησης στο Ουζαμπέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ληφθούν υπόψη από την κυβέρνηση, ιδίως όσον αφορά τον δικαστικό κόσμο και τον κόσμο της δικαιοκορίας. Καταλαβαίνω βέβαια τις ανησυχίες που έχετε για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Τατζικιστάν και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν θα λάβει πλήρως υπόψη τις ανησυχίες αυτές στον διάλογό μας με την εν λόγω χώρα. Όσον αφορά τις οικονομικές ε, μεταρρυθμίσεις, βλέπουμε να υπάρχει πρόοδος, παραδείγματο χάρη, ε, με την υπογραφή ε, ενός μηχανισμού για τη μείωση του χρέους, Πράγμα που θα βοηθήσει μια γεωρική μεταρρύθμιση και θα αντιμετωπιστεί έτσι η ένδια στη χώρα. Οι προσπάθειες αυτές θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε εργασία μας με τον Τζεχισιάν σε πολλές οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ιδιαίτερα τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και φροντίζοντας πλήρη εφαρμογή όλων των μέτρων αυτών οι προσπάθειες μεταρρύθμισης ήδη βασίζονται σε μεγάλο ποσοστό διμερούς ενίσχυσης από την Κομισιόν, 66 εκατομμύρια για την περίοδο 2007-2010, που θα αυξηθεί μάλιστα μέχρι τα 70 εκατομμύρια ε, στα έτη 2011-2013. Ο στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στον ενίσχυση των συγκεκριμένων τομέων, κοινωνική μεταρρύθμιση και ενίσχυση για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Η διαδικασία αυτή θα υποστηριχτεί από την αντιπροσωπεία μας στην Ουτσαμέ και σκοπεύω πριν από τα τέλη αυτού του έτους η περιφερεικά μας εκπροσώπηση εκεί να είναι μια πλήρης αντιπροσωπεία για να ενισχύσει τη διαδικασία μεταρρύθμισης και να φροντίσει σωστή εφαρμογή του PCA και ελπίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να παρακολουθούμε πλήρως την πρόοδο στους κυρίως τομείς, ο οποίος ανέφερα προηγουμένως, και θα τους καταμετρήσουμε έτσι έναντι κάποιων benchmarks που θα έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το λόγο έχει ο εισηγητής κύριος Πέτερλε για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Η απόφαση σύναψη συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των κρατών μελών και του Τατζικιστάν ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη νέα εταιρική σχέση με τις χώρες κεντρική ασία, αλλά και την δέσμευση του Τατζικιστάν ε, να έχει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το εμπόριο και άλλου τομεί. Χαίρομαι που όλα τα κράτη-μέλη επικύρωσαν αυτή τη συμφωνία και μετά το Καζακστάν, την Κυργιζία και το, και το Ουσμπεκιστάν ελπίζω να συναυθεί η παρόμοια συμφωνία και με το Τατζικιστάν. Η ε, Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας που συνήφθη ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες ε, εκπνέει πια. θα πρέπει να εκφράσουμε την, το ενδιαφέρον μας για στρατηγική συνεργασία με το Τατζικιστάν που έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία στην περιοχή. Η σύσπηξη των σχέσεών μας με το Τατζικιστάν θα εξασφαλίσει σταθερότητα, θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, στην εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και θα διασφαλίσει το κράτος δικαίου προσπίζοντας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στο Τζικιστάν συνδέονται κυρίως στη συνδρομή για την καταπολέμηση της φτώχειας, για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, αλλά και την πάταξη της οργανωμένης εγκληματικότητας και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Ε, στην έκθεση περιλαμβάνονται επικρίσεις για το κράτος της δημοκρατικότητας και εκφράσεις ανησυχίες για την οριάζουσα ε, διαφθορά και τα ελληπή κοινωνικά δικαιώματα. Επίσης υπάρχουν ε, μεγάλες αδυναμίες και ελλείψεις στον τομέα της υγείας και της παιδείας. Επ' ευκαιρία της συμφωνίας αυτής εκφράζουμε τις ανησυχίες μας ε, για την χαμηλή τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα την παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών και ελπίζουμε να έχουμε πιο εντατικό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί η πρόοδο στον τομέα αυτό είναι απαραίτητη για την ε, ανάπτυξη των σχέσεών μας. Θα βοηθήσουμε τον Τατζικιστάν να διαμορφώσει ένα σύγχρονο και εύρυθμο κράτος για να διαδραματίσει το ρόλο του στην περιοχή με αποτελεσματικό τρόπο, ιδιαίτερα στην προσπάθεια καταπολέμησης του εξτρεμισμού που εκπορεύεται από το Αφγανιστάν και τις γειτονικές χώρες. Υπάρχουν κάποιες ε, παράγραφοι και για την ενέργεια και για το είδωρ. Η κατάσταση στους τομείς αυτούς ε, ε, έχει σημαντικές συνέπειες για τις ευρύτερες σχέσεις στην περιοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βοήθειά τους και να ευχαριστήσω και την πρεσβεία του Τατζικιστάν για τη στενή συνεργασία. επίση. να ευχαριστήσω θερμά και του συναδέλφου που συνέβαλαν στην έκθεσή μου. Ελπίζω να αναβαθμίσουμε τη μέχρι τώρα σχέση που είχαμε με το Τατζικιστάν και υπό αυτό το πνεύμα ευελπιστώ ότι η συμφωνία αυτή θα, θα εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό. Σα συστήνω λοιπόν θερμά να εγκρίνεται αυτή τη συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία με το Τατζικιστάν. Ευχαριστώ κύριε Πέτελε. Τώρα έχουμε του μετέ γνώμε των πολιτικών ομάδων. Ο κύριο Κασουμαρίκα, εξονομητό τη ομάδα του ΕΕΛΚ. Δημοκράτων. Δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μα τον κύριο Αλόι Πέτερλε, ε, για την ε, πολύ καλή αποουσιαστική άποψη αλλά και πολύ ισορροπημένη έκθεση σε ό,τι αφορά την σύναψη συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τατζικιστάν. Είναι μια χώρα που επικρίνεται συχνά για δημοκρατικό έλλειμμα. Αυτό που, δυστα... που με δυσαρεστεί είναι η έλλειψη ελευθεροτυπία, ανεξεθρησκεία αλλά και η διαφορά. Δεν αφισβητώ τι επικρίσει αυτέ. Θα ήθελα όμω να μην παραβλέψουμε ότι το Τατζικιστάν σημείωσε πρόοδο ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη διαφθορά, τη βελτίωση των σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και σε άλλου ευαίσθητου τομεί. Είναι ένα σχετικά σταθερό κράτο και είναι σημαντικό γιατί κατέχει και στρατηγική θέση στην περιοχή. Αναφέρθηκε πριν από λίγο. Συνορεύει με το Αφγανιστάν και τα συνεφή με αυτό προβλήματα μαζική παραγωγή και λαθρεμπορίου ναρκωτικών, τρομοκρατία και κλιμάκωση του εξτρεμισμού. Μάλιστα συνορεύει και με ένα όλο και ασταθέστερο Πακιστάν. Το Τατζικιστάν μπορεί να γίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση ένας φυσικός σύμμαχος. Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης λοιπόν να συνδράμουμε τη χώρα αυτή στην ολοκλήρωση δημοκρατικής διαδικασίας και να ενισχύσουμε το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό του δυναμικό. Μην ξεχνάμε ότι το Τατζικιστάν είναι η φτωχότερη χώρα από τι πρώην Σοβιετικές δημοκρατίε. Είναι μία από τι 20 μόνο χώρε που περιλήφθηκαν το 2008 στον κατάλογο του ΟΗΕ για τι χώρε που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση των τροφίμων. Χαίρομαι που υπενθυμίζουμε στην έκθεση του Τατζικιστάν του αναπτυξιακού στόχου τη χιλιετία. Δεν θα πρέπει να του ξεχνούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτο εμπορικό εταίρος του Τατζικιστάν και οι δύο πλευρέ λοιπόν θα πρέπει να συμβάλλουν στην άμεση εφαρμογή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης. Πέραν των κριτικών, την πετυχαίνει το Τατζικιστάν, θα πρέπει να στείλουμε και θετικό μήνυμα για να αναπτύξουμε τις επαφές ε, με τη χώρα αυτή και χαίρομαι που η έκθεση του Αλόης Πέτελ δίνει ακριβώς αυτό το μήνυμα. Σας ευχαριστώ εκ μέρου Συμμαχία των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, ο κύριο ε, Ρεϊνάλντι έχει το λόγο. Για ένα λεπτό ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ συνάδελφοι των Τζικιστάν. Ε, αναφέρεται συχνά σε αυτή την αίθουσα. Καλωσορίζουμε όσον αφορά την πλευρά των φιλελευθέρων και δημοκρατών για την Ευρώπη και σαν μέλος τη Επιτροπής ε, διεθνού Εμπορίου για τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Καλωσορίζουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία. Χαιρετίζω και αυτή την απόφαση να προχωρήσουμε με ταχύτητα στην, ε, να γίνει το γραφείο μας εκεί στην περιοχή αντιπροσωπεία. Όπως είπε ο Επίτροπος, κατά τα λοιπά το Τατζικιστάν είναι μια χώρα που μπορεί να εκπλήσει πολύ συχνά καθορίζεται σαν ένα προπύργιο της Ευρώπης. Δεν είναι στην άκρη του κόσμου, αλλά όπως είναι κοντά σε σημαντικές χώρες της Κεντρικής Ασίας, όπω είναι ε, το Αφγανιστάν. Γίνονται σημαντικέ μάχε εκεί για το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών, καταπολέμηση του φονταμενταλισμού, του ολοκληρωτισμού και την παγίωση τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου, που δυστυχώ εκεί είναι πολύ αδύναμοι θεσμοί. Αυτό το με αυτό το μέσο μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα πρόοδου, όχι μόνο εμπορικά αλλά και πολιτικά και πολιτισμικά βήματα πρόοδου. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Τώρα για τους πρασίνους είχε η κυρία Χάουταλα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Τατζικιστάν πλη... Ε, ε, πλησίασε περισσότερε συνθήκε για του όρου για την υπογραφή τη συμφωνία από ότι το Σμπεκιστάν και το Τουρκμενιστάν όπου εκεί σοβεί η δικτατορία. Το Τατζικιστάν είναι σε καλύτερη θέση και επηρέασε τα τεκτενόμενα Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη χώρα και θα τα επηρεάσει περισσότερο χάρη σε αυτή τη συμφωνία. Και σε αυτή τη συνεργασία θα επικεντρωθούμε στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη δημοκρατία και θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το κράτος δικαίου. Και είναι ικανοποιητικό που ακούσαμε ότι στο Τατζικιστάν υπάρχει και θέση διαμεσολαβητού αυτό είναι σημαντικό βήμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει πλήρω αυτό το νέο θεσμό του διαμεσολαβητή, του συνηγόρου του πολίτη. Ε, επιτρέψτε μου να επανέλθω στο θέμα των υδατίνων αποθεμάτων. Αυτή η χώρα έχει σημαντικά αποθέματα ύδατο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει το Τατζικιστάν να εκμεταλλευτεί καλύτερα το νερό του με βιώσιμο και δημοκρατικό τρόπο, λαμβάνοντα υπόψη τα συμφέροντα και των χωρών που είναι ε, κατάντι των υδάτων αυτών και ίσως ε, να, ε, εάν κατασκευάσουν φράγματα στο Τζικιστάν, να έχουν δυσάστη συνέπειε σε άλλε χώρε. Οι πράσινοι δίνουν σημασία σε μη περιφερειακή συνεργασία, ούτω ώστε η οικονομία αυτών των χωρών να μπορέσει να προωθηθεί. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κ. Τάνοκ, μέρο του κόμματο, το έχει Ευχαριστώ. Το Τζικιστάν δεν έχει ενέργεια και ε, ρηκτό πλούτο όπω άλλε χώρε τη Κεντρική Ασία, όμω αυτό δεν είναι δικαιολογία για περιθυριοποίηση του Τατζικιστάν Ει βάρο των, εν συγκρίση με πιο πλούσιους γείτονε. Η Κεντρική Ασία είναι μια περιοχή που είναι ζωτική για την πολιτική και ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ενισχυθούν οι σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιε χώρε προχωρούν πιο γρήγορα από άλλε. Αυτό είναι ανεπόφευκτο, αλλά θα πρέπει να συλλογικά να δεσμευτούμε προσπαθώντα να βελτιώσουμε του δεσμού με περιοχή που ήταν διπλωματικά απομονωμένη και ξεχασμένη, κυρίω από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζοντα κάποιε χώρε Κεντρική Ασία έναντι άλλων, ίσω δημιουργήσει διαφορά και διέρεση στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, οι Ισλαμιστέ τρομοκράτε περιοχή έδειξαν αποφασιστικότητα να εκμεταλλευτούν τη φτώχεια και ανεπαρκή διακυβέρνηση, ούτω ώστε να κάνουν πιο ριζοσπαστικού του κατοίκου και να σπείρουν το μίσο. Η κυβέρνηση του Τατζικιστάν απέρριψε τον εξτρεμισμό και με τη βοήθεια τη διεθνού κοινότητα επιδιώκει τώρα να εδραιώσει την δημοκρατία. Το Τατζικιστάν εξακολουθεί να έχει τα σημάδια ενό εμφυλίου πολέμου μεταξύ των υπασπιστών του Τζιχάτ και των κοσμικών δυνάμεων μετά την ε, κατάρρευση τη Σοβιετικής Ένωση τη δεκαετία των 90. Ο το Τατζικιστάν δεν θέλει να επιστρέψει η αιματοχυσία και γι' αυτό με γενναιότερη υποστήριξαν τι επιχειρήσει του ΝΑΤΟ κατά του, των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Η αποστολή ISAF στο Αφγανιστάν είναι ζωτική σημασία για το Τατζικιστάν και για το μέλλον τη χώρα και την προσπάθεια που καταβάλει να βρει στη Δύση μια άγκυρα ασφαλείας. Ο εκδημοκρατισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Τατζικιστάν είναι στο τομέα ατελή. Αλλά βεβαίω διάλογο και προσπάθεια πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα ενθαρρύνει το Τατζικιστάν για να επιφέρει θετικέ αλλαγέ. Σίγουρα αυτή είναι η άποψη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω όσον αφορά τη Λευκορωσία και το Ουσμπεκιστάν. Το Τατζικιστάν λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί παρομοίω. Η ομάδα ICR υποστηρίζει ε, βαθύτε στρατηγική πολιτική οικονομική συνεργασία με το Τατζικιστάν βάσει δεσμεύσεω προ πρόοδο, άνοιγμα, δημοκρατία και υψηλέ προδιαγραφέ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοκ. Και τώρα. Εκ μέρου τη ΓΚΟΕ το λόγο έχει η κυρία Λέζινγκ για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σε μία συνάντηση που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συζητήσαμε για το ρόλο που θα διαδραματίσει η συμφωνία αυτή σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μου είπε απερίφραστα ότι μετά τη θέση ισχύ της συμφωνίας αυτής σίγουρα θα συσφιχθούν οι σχέσεις ε, με την υπηρεσία Frontex και οι διαδικασίες επαναπροώθησης ε, προς το Αφγανιστάν θα διευκολυνθούν. Έγινε πολλής λόγος για το μήκος ε, των συνόρων του Τατζικιστάν με το Αφγανιστάν. Η συμφωνία αυτή λοιπόν θα αποτελέσει ένα επιπλέον μέτρο για να εξασφαλίσει την καταπίεση των μεταναστών στην Ευρώπη. Διαπιστώνουμε ότι αυτή η καταπολέμηση της μετανάστευσης έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής μας πολιτικής. Και μάλιστα έχουμε καταγγείλει πολλάκις ε, τις ε, απάνθρωπες συνθήκες τις οποίες διαβιούν οι μετανάστες σε πολλές χώρες, για παράδειγμα στην Ουκρανία. Και τέτοιου είδους συμφωνίες επιδεινώνουν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και μάλιστα παραβιάζουν τη συνθήκη της Γενέβης, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων αυτών. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με το ουσιαστικό πρόβλημα και να μην καταπιέζει και να μεταχειρίζεται τους μετανάστες. Για μας είναι ακατάλληλη αυτή η έκθεση και την αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερο σκεπτικισμό. Το λόγο έχει εκ μέρους του ΙΕΒΔΕ ο κύριος Μπέλντερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή μου δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα. Αφενός Χαίρομαι που ο κύριος Πέτρελε στην πρόταση ψηφίσματος του εντοπίζει μερικά ευαίσθητα σημεία και τομείς στην τατζικική κοινωνία. Βέβαια, μιλούμε ε, κατεφημισμό για το Τατζικιστάν, αποκαλώντας το σταθερό κράτος. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρησιμοποιούνται τέτοιες εφημιστικές δηλώσεις. Γιατί έχουν επαγγελθεί πολλές κατηγορίες κατά το Τατζικιστάν. Η παράγραφος 2 μιλά για την απογοήτευση των τατζικικών αρχών. Εγώ θα προτιμούσα να μιλούμε για την απογοήτευση της προτεσταντικής μειονότητας, γιατί ο θρησκευτικό νόμο παραβίασε στοιχειώδεις θρησκευτικέ ελευθερίε των κοινότητων αυτών. Και αντί για απογοήτευση των τατζικικών αρχών, θα πρέπει να ζητήσουμε από τι αρχέ αυτέ να τακτοποιήσουν πρώτα τα του οίκου του πριν προβούν σε Σας ευχαριστώ κύριε Μπέλτερ. Ο κύριος Αρλάκη έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Είμαι υπέρ της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με το Τατζικιστάν. Πιστεύω ότι συμβάλλει στην πρόοδο και προωθεί τη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και Τατζικιστάν. Η χώρα αυτή είναι πολύ σημαντική για πολλού και διάφορου λόγου. Θα περιοριστώ στην αναφορά ενό μόνο, στη συμβολή, στη σταθερότητα και την ασφάλεια τη υπήρου μα. Το Τατζικιστάν βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι λαθρεμπορίου ναρκωτικών από το Αφγανιστάν προ την Ευρώπη. Είναι χώρα διέλευση. Τουλάχιστον 30% τη ηρωίνη που παράγεται στο Αφγανιστάν μπαίνει, στη, ε, μπαίνει στην ε, Ευρώπη και τη Ρωσία μέσω του Τατζικιστάν. Η διεθνή κοινότητα ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια μια σημαντική προσπάθεια στο Τατζικιστάν, ενισχύοντα τα διάφορα συστήματα και προγράμματα ελέγχου των ναρκωτικών. Και βλέπουμε ικανοποίηση μια δεκαετία μετά ότι το σύστημα λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Πρόκειται για μια άμεση συμβολή στη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης η σύναψη αυτή τη συμφωνία με το Τατζικιστάν. Βέβαια, αδυναμίε υπάρχουν ακόμη και πολλοί συνάδελφοι υπογράμμισαν τα προβλήματα που μαστίζουν το Τατζικιστάν σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ένδια και ούτω καθεξής. Πάντως, ε, αυτή η συμφωνία είναι ό,τι καλύτερα μπορεί να κάνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και είμαι αναφανδόν υπέρ της συμφωνίας. Καλώς κύριε Αρλάκη. Ξέρουμε ότι ένα λεπτό είναι ελάχιστος χρόνος. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα σε ένα γύρο της διαδικασίας ΚΑΤΣΙΔΙΑΗ για πέντε λεπτά. Πρώτος έχει στήσει ο κ. Παντσέρη. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω και εγώ ότι πραγματικά είναι άκρο θετική αυτή η συμφωνία συνεργασίας με το Τατζικιστάν και βοηθά να πετύχουμε κάποιους στόχους που θεωρώ σημαντικούς και είναι συγκεκριμένοι. Πρώτος στόχος αφορά τη στρατηγική θέση της χώρας που μπορεί πραγματικά να είναι χρήσιμη για να ευνοήσει μια δημιουργία μιας περιοχής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας. Δεύτερος στόχος είναι να ευνοηθεί ανάπτυξη της χώρας οικονομικά και κοινωνικά να αναπτυχθεί, διότι ξέρουμε ότι είναι η μία χώρα από τις στοχότητες περιοχής. Και τέλος, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να φροντίσουμε τους ώστε ελευθερία, δημοκρατία και δικαιώματα να είναι τα θεμελιώδη στοιχεία που θα πρέπει να καθοδηγούν την εφαρμογή της ε, συμφωνίας. Πέρα από τα όρια που μπορούν να αντιμετωπιστούν, εγώ νομίζω ότι χαιρετίζουμε θετικά ε, αυτό το μέτρο και θα το ψηφίσουμε στην ε, Ολομέλεια. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κύριος Κάτσε έχει το λόγο. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Αλόης Πέτερλε για την καταπληκτική του έκθεση. Σταν σημαίνει κράτος και το Τατζικιστάν είναι το τελευταίο κράτος ε, που το όνομά του τελειώνει σε Σταν και που μέχρι τώρα δεν είχε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ήταν αδικία. Η σταθερότητα στην περιοχή αυτή είναι προς το συμφέρον όλων μας είναι και προς το στρατηγικό συμφέρον ολόκληρου του κόσμου. Γιατί οι χώρες αυτές έχουν σημαντική θέση και λειτουργούν ως όχημα σταθερότητας. Οι προσπάθειές μας λοιπόν θα πρέπει να κατευθύνονται προς όλες τις ε, χώρες της περιοχής, άσχετα με τις διαστάσεις τους και άσχετα με τους ενεργειακούς τους πόρους και τον ορυκτό τους πλούτο. Γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ θερμά και τον εισηγητή αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Επίτροπο και τη Σουηδική Προεδρία γιατί κατάφεραν να καλύψουν αυτό το κενό ε, που ανήκει πια στο παρελθόν. Το μέλλον θα είναι λαμπρότερο. Ευχαριστώ. κύριο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Να θέσω μια ερώτηση πολύ καλώς προτάθηκε η σύναψη της συμφωνίας αυτής τη εταιρική σχέση και συνεργασίες. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά έχω μία ερώτηση προς την Υπουργό Μάλμστρεμ. Στις διάφορες δραστηριότητες που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση βοηθώντας το Τατζικιστάν να καταρτήσει καλύτερα και να επιμορφώσει τους φύλακες ε, και τους αρμόδιους με τη διαχείριση των συνόρων στο Αφγανιστάν. Γιατί τα σύνορα αυτά έχουν μήκος 1500 χιλιόμετρα ε, και το Τατζικιστάν έχει πολύ σοβαρά προβλήματα με τον έλεγχο αυτών των σύνορων. Πολλό δε μάλλον που υπάρχει και η αφγανική μειονότητα. Θα Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση το, το Τατζικιστάν, δηλαδή να παράσχουμε συνδρομή στην επιμόρφωση και κατάρτιση των φυλάκων που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των συνόρων με το Αφγανιστάν. Ευχαριστώ συνάδελφε. Δεν βλέπω κανέναν. Είχατε ζήσει το λόγο για το Καστιάι, συνάδελφε. Όχι. Ο κύριο Πάσελτ όμως, από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι, εκεί πίσω. <clears throat> Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια θαυμάσια έκθεση αυτή που προτιμούσε ο συνάδελφο Πέτερλε. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι αυτές οι χώρες που αγαπούν την ελευθερία στην Κεντρική Ασία είναι η σημαντικότερη εταίροι μας. Αυτή η περιοχή πολλές φορές ελέγχεται από ηγετικέ δυνάμεις. Εδώ και χιλιαετίες για πρώτη φορά είναι πάλι ελεύθερη και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε με εταιρική σχέση ελευθέρων. Προηγουμένω κάτι άκουσα για εγκληματικότητα. Βέβαια, πρέπει από κοινού να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα. Αλλά θα πρέπει καταρχήν να δούμε τον πολιτισμό των χώρων αυτών και να δούμε ότι πρόκειται για παμπάλιε εμπορικέ ε, χώρε, όπου δεν είχαν εμπόριο μόνο με ε, ναρκωτικά, αλλά με προϊόντα που ήταν σημαντικά και για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Να πούμε λοιπόν ότι πρόκειται για ε, για εταιρική σχέση και όχι αίγεση. Ευχαριστώ κύριε Πόσελ, πρόεδρος. Τελευταίον, είδα τον κύριο Πλεύρη που ζητούσε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στο θέμα της εγκληματικότητας που αναφέρθηκε όπως επίσης και της λαθρομετανάστευσης. Είναι γεγονό ότι το Τακιστάν βρίσκεται σε ένα νευραλγικό σημείο, σε μια γεωπολιτική θέση που θα πρέπει να εξετάσει η Ευρώπη πώ θα καταφέρουμε να περιορίσουμε αφενός την εγκληματικότητα η οποία παρατηρείται ειδικά στα ναρκωτικά από το αφγανιστάν αλλά πρωτίστως τις μεταναστευτικές ροές. είναι γεγονός ότι πλέον η ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη μεταναστευτική ροή από το αφγανιστάν μέσω του τατζικιστάν και από τις άλλες χώρες πράγμα που σήμερα το πληρώνουν πρωτίστως οι μεσογειακές χώρες ε, μάλτα κύπρος ελλάδα ιταλία αλλά αργότερα είναι με μαθηματική ακρίβεια ότι θα το ε, πληρώσουν και όλες οι χώρες της βόρειας ευρώπης. πρέπει οπωσδήποτε να σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων αυτών των ανθρώπων που έρχονται από εκείνες τις χώρες αλλά κάποια στιγμή και η ευρώπη πρέπει να κατοχυρωθεί και να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε όλη αυτή τη μεταναστευτική ροή από την ασία έχοντας ακούσει τους μελητές του Κοινοβουλίου και τον εισηγητή, το λόγο έχει η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Όπως είπε ο κύριος Πέτερλε στην έξοχη αναφορά του, η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσεως και Συνεργασίας είναι ένα κομμάτι μιας μεγαλύτερης στρατηγική για αυξημένη ασφάλεια και σταθερότητα στην Κεντρική Ασία. Και βέβαια πρέπει να δούμε τη γενικότερη εικόνα, διότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα βαθιά ριζωμένα που πλήττουν πολλές χώρες, ανάμεσα στι οποίε Πακιστάν, Αφγανιστάν. Η κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητες τη, τα χαρακτηριστικά τη, τα προβλήματά τη. Και αυτό το συμπεριλαμβάνει ο κ. Πέτερλε με συστηματικό τρόπο στην έκθεσή του. Χαίρομαι όλο ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να υψώνει το φλάμπουρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κατά Είναι ένα πρόβλημα στο Αφγανιστάν. Απομένουν πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Γι' αυτό είναι τόσο χρήσιμο, όπω είπε η Επίτροπο, να έχουμε αυτό το διάλογο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και είμαι σίγουρη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη φορά θα είναι πολύ ξεκάθαρη όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες και τι προσδοκίες έχουμε έναντι του Τατζικιστάν. Έγινε και μια διάσκεψη που στηρίξαμε τον Ιούλιο πάνω σε αυτό το θέμα όπου στόχο είχε να ενισχυθεί το κάτω δικαίου στο Τατζικιστάν. Υπήρχαν εκπρόσωποι της κοινωνία των πολιτών, διαφόρων οργανώσεων, ε, ειδικοί για εξωτερικά θέματα, καθώς και πολλοί άνθρωποι από τις αρχές του Τατζικιστάν, πολλοί πρόσωποι των αρχών του Τατζικιστάν. Ε, θέλαμε να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, το κράτος δικαίου ε, και είναι και το θέμα των υδάτων. Εξαιρετικά σημαντικό θέμα για την περιοχή και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει βιώσιμα προγράμματα για παραγωγή υδροελεκτρική ενέργεια. Αυτά τα προγράμματα, αυτά τα έργα βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες, θα πρέπει να έχουν μια περιφερειακή προοπτική και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ε, ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής. Ο κύριος Στέμκα αναφέρθηκε στη διαχείριση των συνόρων. Είναι σημαντικότατο ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει 66 εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή μέχρι το 2010 και 17 εκατομμύρια την επόμενη τριετία. 70 εκατομμύρια. Και πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ενισχυθούν οι έλεγχοι των συνόρων και η εκπαίδευση του προσωπικού του αρμοδίου. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανέλθει όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Κυρία Πρόεδρε, συνοψίζοντας, υπάρχουν πολλά δύσκολα προβλήματα στο Τατζικιστάν και στην υπόλοιπη περιοχή αλλά υπάρχει ελπίδα. Δεν πρέπει να υποτιμούμε όμως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Χαίρομαι που υπάρχει συνένεση από ό,τι βλέπω στο Κοινοβούλιο Δηλαδή θεωρείτε και εσείς σημαντικό να κάνουμε το βήμα προς τη Συμφωνία Συνεργασίας και εταιρική Σχέσης. Θα έχουμε έτσι ένα καλύτερο εργαλείο στα χέρια μας για να εργαστούμε για καλύτερη σταθερότητα και να επιλύσουμε τα προβλήματα και να επιδιώξουμε ένα διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη δημοκρατία με αυτή τη χώρα. Αποτελεί ένα σημαντικότατο βήμα προόδου και καλύπτει ένα κενό που υπήρχε σε αυτή την περιφερειακή στρατηγική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει πάλι εξ ονόματο τη Επιτροπή η Επιτροπή κυρία Φεραίρο Βάρντερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. <clears throat> Καταρχήν, ε, επιτρέψτε μου να πω ότι βέβαια εδώ και πολύ καιρό πιστεύουμε ότι μια θετική Ευρωπαϊκή Ένωση Κεντρική Ασία είναι πάρα πολύ σημαντική και ότι θα έχει πραγματικά θετικέ επιπτώσει στην ασφαλή, σταθερότητα και στην ευμάρεια των διαφόρων χωρών τη Κεντρική Ασία. Όπω δικαίω είπε ο κ. Στένοκ, δεν θα πρέπει να περιθωροποιήσουμε το Τατζικιστάν Τον Αντίος θα πρέπει νομίζω με αυτή την τόσο φτωχή χώρα της Κεντρικής Αμερικής, ε, ε, θα πρέπει να αναπτύξουμε σχέσεις. Ε, παραδέχομαι ότι υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις για τη χώρα αυτή. Ο κ. Σαλάκη ανέφερε ότι το Αφγανιστάν παραμένει η κύρια χώρα παραγωγής ηρωίνης του κόσμου και κινείται το ναρκωτικό αυτό μέσω του Τατζικιστάν. Το όπιο και, το... <clears throat> και η περνάνε από τον, ε, το Ιράν και το Πακιστάν στο νότο αλλά και από το Τατζικιστάν, το Μεγκιστάν και άλλες χώρες στο Βορρά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Παρ' αυτό όμως αναγνωρίζουμε ότι η παραγωγή ναρκωτικών έχει μειωθεί στο Αφγανιστάν. Και τώρα θα πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να αυξήσουμε αυτή την τάση της μείωσης. Επίσης έχει εισαχθεί ένα σύστημα διαχείρισης των συνόρων που καταπολεμά το λαθρεμπόριο και επιτρέπει τις χώρες αυτές όμως να αναπτύξουν ε, ένομο εμπόριο και είναι κατά της παραγωγής ναρκωτικών. αυτά τα θεσμικά όργανα που έχουμε δημιουργήσει λειτουργούν πολύ καλά και εμείς εκπαιδεύουμε, εκπαιδεύουμε τα άτομα εκεί. Ε, είναι και αυτό ένα τμήμα του προγραμματός μας. Όσον αφορά τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιτρέψτε να σα πω δύο λόγια. Πράγματι, η νόη συμφωνία εταιρικής σχέση και συνεργασία θα μας δώσει μια δυνατότητα να εμβαθύνουμε το διάλογό μας με το Τατζικιστάν στον τομέα αυτό. Υπάρχει αυτή η ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε με τις αρχές ε, του Τατζικιστάν όλα τα σχετικά θέματα, τα <clears throat> δικαιώματα των γυναικών και την θρησκεία, κύριε Μπέλλερ, ακριβώς επειδή υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί. Το νερό αναφέρθηκε επίσης και θα ήθελα να σας πω ότι εδώ και πολλά πολλά χρόνια εγώ γνωρίζω αυτό το πρόβλημα και προσπάθησα να, να βοηθήσουμε τους ε, Τατζίκους και τώρα εμείς ε, παίρνουμε, ε, παίζουν, τους δίνουμε δυνατόν να παίξουν ένα ρόλο διευκόλυνση μεταξύ των διαφόρων χωρών της Κεντρικής Ασίας. Θα πρέπει νομίζω αυτό να λάβει χώρα σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και το Τσίχης το και από την άλλη μεριά το Ουσπεκιστάν, το Τουρκμεκιστάν και μόνο εάν ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι χώρες θα είναι προς όφελος όλων οι εξελίξεις το έχουμε αυτό υπόψη μου και μέσα στα πλαίσια αυτά υπάρχει τώρα ένας εθνικός ε, διάλογος πολιτικής για τα ΕΟΙΔΟΡ όπου θα εξεταστούν όλα αυτά τα θέματα. Και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Τελειώνοντας, Πρόεδρε, έχω να πω ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να υποστηριχθεί το τελευταίο ε, βήμα για την επικύρωση της Συμφωνίας Τερικής και Συνεργασίας. Ε, όλα αυτά προς όφελος των πολιτών. Θα αποστείλουμε ένα θετικό μήνυμα προς το Τατζικιστάν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τις ε, υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε στα πλαίσια δικής μας για την Κεντρική Ασία και αυτό θα οδηγήσει σε μια εταιρική σχέση σημαντική για τη δική μας ασφάλεια και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη περιφερειακή συνεργασία που είναι τόσο σημαντική για την σταθερότητα της Κεντρικής Ασίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το λόγο έχει τώρα για μια φορά ο εισηγητή, κύριο Πέτελε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σεσίλια για τα ευγενικά της λόγια, για το φως που έχει στην υπόθεση, της νέες διευκρινήσεις που μας έκανε. Όλα αυτά δείχνουν ε, μια μεγαλύτερη ομόνοια και σύντοση απόψεων προ προς το θέμα αυτό μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και την ανάγκη μιας σύσφυξης των σχέσεων και μιας ε, πάγιας συνεργασία με το Τατζικιστάν λόγω του ιδιαίτερου ρόλου που διαδραματίζει στην περιοχή. Και ελπίζω ότι το Τατζικιστάν ε, θα δείξει ιδιαίτερη πυγμή και προσήλωση και στην εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, όσοι έδειξε και για την σύναψή της. Θα πρέπει και εμείς να παρακολουθήσουμε ε, μέσω των αντιπρο... της αντιπροσωπείας μας για τις επαφές με την Κεντρική Ασία να μεριμνήσουμε για την σωστή εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Αύριο μάλιστα θα υπογραφεί και τελική πράξη της συμφωνίας. Ευελπιστώ ότι θα συγκεντρωθεί ε, συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της συμφωνίας αυτής και μετά τη θέση ισχύ της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Τατζικιστάν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη και διμερή αλλά και πολυμερή συνεργασία με τη χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σίτα. Έχω λάβει ένα ψήφισμα μια πρόταση ψηφίσματο σε Επιτροπή για Εξωτερικά Θέματα. Κλείνει η συζήτηση εδώ. Η ψηφορία για την πρόταση ψηφίσματο θα λάβει χώρα αύριο.